θανατικής ποινής. Εδώ και δεκαετίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ της κατάργησης θανατικής ποινής σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι είναι πεπισμένοι πως όσο φρικτά και αν είναι τα εγκλήματα κάποιου δεν επιτρέπεται να υπάρξει άλλη μία δολοφονία. Μόνο πέρσι σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία δολοφονήθηκαν 682 άνθρωποι σε 21 χώρες και πιθανώς υπάρχουν και άλλες χιλιάδες εκτελέσεις που δεν ε, επιβεβαιώνονται επισήμως. Επίσης και το 2012 η Κίνα, το Ιράν, το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελεστέντων παγκοσμίω παραμένουν 23.000 άνθρωποι φυλακισμένοι και αναμένουν την εκτέλεσή τους. 1.700 καταδίκες σε θάνατο υπήρξαν το 2012. Λυπούμεθα για το ότι χώρες όπως η Γάμβια, η Ινδία, η Ιαπωνία και το Πακιστάν επα... ξανάρχισαν να εκτελούν ανθρώπους το 2012. Αλλά Υπάρχουν και καλές ειδήσει. Ο αριθμός των αντιπάλων της θανατικής ποινής αυξάνεται. Σε 97 χώρες έχει καταργηθεί η θανατική ποινή. Σε 140 χώρες κυβερνήσεις και κοινοβούλια έχουν εκφραστεί κατά της θανατικής ποινής. Οπωσδήποτε αξιοσημείωτες είναι οι εξελίξεις της ΕΠΑ. Ένα τρίτο των πολιτιών έχουν αποφασίσει να καταργήσουν θανατική ποινή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώ πως κατά συντριπτική πλειοψηφία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να στηρίξει αυτές τις θετικές εξελίξεις. Και θα ήθελα εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσω να καταργηθεί επιτέλους αυτή η απάνθρωπη ποινή. Ich Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος πρώτος. Ευχαριστώ. Το προσπεράσατε, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη από όλες τις πολιτικές ομάδες που στήριξαν την πρότασή μου για την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ στη Μαλάλα Σαυσάη. Είναι καταπληκτική η δράση αυτής της εφήβου ε, και ο διορισμός αυτός ε, ε, έγινε δεκτός από τις πολιτικές ομάδες γιατί το επιχείρημά της ότι και τα νέα κορίτσια έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση χρήζει αμέριστης υποστήριξης και είμαι ευγνώμων προς τη διάσκεψη των Προέδρων ε, που την, έκρινε ως κατάλληλη για το βραβείο Ζαχάροπ γιατί θα γίνει ίνδαλμα και πολλών άλλων κοριτσιών που έχουν δικαίωμα στην παιδεία. Κύριε Βάτσον, δεν ξέρω κατά πόσον ήταν διαδικαστικό αυτό. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κινηθείτε εντός του κανονισμού. Επί της διαδικασίας, κύριε Γκόμες, αλλά επί της διαδικασίας όμως. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ε, πολύ ανησυχητικέ ειδήσει που παίρνουμε από την Λιβύη για την απαγωγή του Πρωθυπουργού Αλίζη Ντάν από μια ένοπλη ομάδα σήμερα το πρωί. Ευτυχώς μάθαμε ότι απελευθερώθηκε τελικά, αλλά αυτό δείχνει πόσο λεπτή είναι η κατάσταση στη Λιβύη και πόσο τεράστιε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Εγώ, ω μόνιμη συγγήτρια για το θέμα αυτό, πέρασα το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λιβύη με την κυρία Νατάλια Χαφαλόβα, την επικεφαλή αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι είναι η στιγμή αυτή για να εκφράσουμε την ελεγγύη μα προ όλου όσους προς όλους ε, ε, στη Λιβύη προσβλέπουν σε ένα δημοκρατικό μέλλον και το κράτος δικαίου. Σας ευχαριστώ Κύριε Γκόμες, καταλάβαμε αυτό που θέλατε να πείτε, αλλά ε, ούτε και αυτό δεν ήταν επί της διαδικασίας. Γι' αυτό, συνάδελφοι, σας ανακοινώνω. Δεν είναι δυνατόν πολιτικές ανακοινώσεις να βαφτίζονται παρεμβάσεις επί της διαδικασίας. Είναι κατάχρηση. Αυτό όσο και αν έχω κατανόηση ως πολιτικός για το μήνυμα που θέλετε να περάσετε, σας παρακαλώ να μείνουμε στα πλαίσια της συζήτησης της διαδικασίας. Κυρία Σινκλέρ, ναι, έχετε το λόγο κυρία Σινκλέρ. Thank Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως διαδικαστικό. Πρέπει να πούμε ότι εκπροσωπώντας τα West Midlands ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο, και όπου έχουμε στο Queen Elizabeth νοσοκομείο στο Birmingham μια πολύ νεαρή γυναίκα η οποία πραγματικά θα άξιζε το βραβείο αυτό. Αυτό που θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε, είναι ότι είναι πάρα πολύ απογοτευτικό το ότι ουσιαστικά δεν δείξατε σεβασμό απέναντι στην Ολομέλεια και ότι Ανακοινώθηκε πρώτα στο Twitter αυτό, πριν από 30 λεπτά. Νομίζω λοιπόν ότι δεν δείξατε τον δέοντα σεβασμό απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνοντα την ανακοίνωση για τον βράβευση τη Μαλάλα πριν από 30 λεπτά στο Twitter πρώτα και όχι εδώ, στο Κοινοβούλιο. είπα στην διάσκεψη των Προέδρων, μπορείτε να το δείτε στα πρακτικά, πως μετά της, τη λήψη της απόφασης ρώτησα τους συναδέλφους εάν θέλουν ε, να το ανακοινώσουν στο Twitter. Προφανώς συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς περιφρόνησα έτσι το... την Ολομέλεια. Δεν θεωρώ ότι με την ανακοίνωση μιας τέτοιας απόφασης περιφρόνησε την Ολομέλεια και δεν, δεν νομίζω να χρειάζονταν να κρατηθεί μυστική μια τέτοια απόφαση. Δεν έχω κάποιον άλλο τέτοιο λόγο. Α, κύριε Μοργκάτη. Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια τη χρεθνή συζήτηση για την κατάσταση των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη δική μου παρέμβαση, ο κύριος Φραγκάγγελ από το ΕΛΚΑ είπε ότι εγώ λέω ψέματα, ότι ψεύδομαι επειδή ουσιαστικά σας ενημέρωσα για το τι γίνεται στην Ιταλία όσον αφορά τους ε, Ρωμά, πράγματα ιδιαίτερα γνωστά, άλλωστε έχουν απασχολήσει και τις εφημερίδες. Δεν μου δόθηκε δυνατότητα να απαντήσω, ότι ο κύριος Έγγελ χρησιμοποίησε την μπλε κάρτα. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να ζητήσει επισήμως συγνώμη ο συνάδελφος αυτός από μένα και ουσιαστικά νομίζω ότι θα έπρεπε σε διαφορετική περίπτωση να επιβληθούν κάποιες κυρώσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, ποτέ δεν δικαιολογεί το άνθρωπος αυτός να απευθύνεται σε μένα λέγοντας ότι εγώ ψεύδομαι. Κάνω, κάνω την εξή πρόταση. Θα δούμε τα πρακτικά και εάν θεωρείτε παράδεκτη την συμπεριφορά του κυρίου Έγγελ θα ε, ζητήσω τον κύριο Έγγελ να πει πως δεν είναι δυνατόν να σας ε, λέει ψεύτη. Ε, υπό την προϋπόθεση ότι θα δούμε τα πρακτικά σας ευχαριστώ. Δεν ζητάει κάποιος άλλος τον λόγο. Την Προεδρία αναλαμβάνει ο κύριος Κάρας. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στην ε, ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την έκθεση Knights Utenbrook.